die gibt dan in principe kan ik met the base camp. Ladies and gentlemen. Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα να αρχίσουμε παρακαλώ. Λόγω υλικοτεχνικών προβλημάτων έχουμε μια μικρή καθυστέρηση. Ε, θα ήθελα να κάνω πιο σύντομα τα εισαγωγικά μου σχόλια για να κερδίσουμε χρόνο. Ε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διοργανώνει το σημερινό σεμινάριο κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου με τη συνεργασία του Τμήματος Περιπολιτικών του Κοινοβουλίου Ε, δεν είναι ακριβώς βέβαια εργαστήριο, πρόκειται για μια στρογγυλή τράπεζα υψηλού επίπεδου. Στα αριστερά μου έχουμε τον Επίτροπο, κύριο Ντεγκούχτο, για θέματα εμπορίου. Τον Υπουργό παρά τον Πρωθυπουργό της ε, Ουκρανίας. Πρόκειται για μια συνεδρίαση υψηλού επίπεδου. Η διμερή σχέση με την Ουκρανία τα πρόσφατα χρόνια αποτέλεσε ένα από τα κεντρικά ζητήματα της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και από τότε που θεσπίστηκε η Ανατολική Εταιρική Σχέση το 2009, η Επιτροπή ΙΝΤΑ διαπίστωσε πόσο σημαντικά θα ήταν ε, τα εμπορικά και οικονομικά ζητήματα στα πλαίσια της ε, συμφωνίας ε, σύνδεσης με την Ουκρανία και εντόπισε το δυναμικό για να διευρύνει τις εμπορικές αυτές σχέσεις. Παρακολουθήσαμε ως εκ τούτου εκ του σύνεγγυς της διαπραγματεύσης... για τη σύναψη μίας εις βάθους και σφαιρικής συμφωνίας ελευθέρων εμπορικών συναλλαγών που είναι και το αντικείμενο της σημερινής μας συνεδρίασης. Έχουμε ένα μόνιμο εισηγητή στην Επιτροπή μας, τον κύριο Παβεζαλεύσκη, αυτό το θέμα εδώ στα δεξιά μου από το ΕΛΚ που επίσης ε, είναι αντιπρόεδρος της Επιτροπής Ίντα του Κοινοβουλίου. Θα συμφωνήσει μαζί μου ότι η σύναψη αυτής της σφαιρικής και σε βάθος εμπορικής συμφωνίας ενισχύει την πορεία της Ουκρανίας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα οδηγήσει σε μεγαλύτερη ολοκλήρωση, θα είναι υποφελής για τις επιχειρήσεις και εν τέλει θα ενθαρρύνει την Ουκρανία ώστε να συνεχίσει ε, τις ε, θεσμικές ε, μεταρρυθμίσεις που διεξάγει για να εγκατασταθεί το κράτος δικαίου και ε, να βελτιωθεί το επιχειρηματικό κλίμα. Είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντικό να εξετάσουμε τις επιπτώσεις μιας τέτοιας συμφωνίας ε, και επιχαίρω γιατί έχουμε εδώ αξι... τους αξιότιμους βουλευτές που θα συμμετάσχουν στις εργασίες μας. Ε, τις τελευταίες εβδομάδες ε, βλέπουμε δύο εξέχουσες φυσιογνωμίες που συμμετείχαν στις διαπραγματεύσεις ο Επίτροπος κ. Δεγκούχτο και ο κ. Άντρι Κρουιγεφ, ο Υπουργός Πρωθυπουργός στην Ουκρανία που είναι αρμόδιος για την τα θέματα εμπορίου και την οικονομική ανάπτυξη. Σας ευχαριστούμε που ήρθατε. Ξέρετε ότι η σχέση με την Ουκρανία ε, συνιστά ε, προτεραιότητα και για την ε, τωρινή Προεδρία του Συμβουλίου. ορίζουμε, λοιπόν τον κύριο Μάρτιν Κορολέτσε που είναι υφυπουργό στο Υπουργείο Οικονομικών της Πολωνίας. Ευχαριστούμε για την παρουσία σας. Τέλος, ο τελευταίος προσκεκλημένος μας είναι ένας επιφανής Πολωνός καθηγητής, πρώην βουλευτής στην στο Κοινοβούλιο της Πολωνίας και ειδικό οικονομικά θέματα είναι ο Δ. Μάρεκ Νταμπρόφσκι. Ε, θα, μας, ε, θα συμμετάσχει με την τεχνογνωσία του ε, στην σημερινή συζήτηση. Θα θέλαμε να η σημερινή συζήτηση να διεξαχθεί σε δύο στάδια. Πρώτον θα ακούσουμε τα μέλη του πάνελ, κατόπιν θα ακολουθήσει η συζήτηση και στο δεύτερο τμήμα της συζήτησης θα ακούσουμε την παρουσίαση από τον ε, εμπειρογνώμονά μας, τον ε, δόκτωρα Νταμπρόσκι και θα συνεχίσουμε με έρωτα απαντήσεις ε, όπου θα συμμετάσχει ο κύριος Ντότορ που είναι υποδιευθυντής του αντίστοιχου τμήματος στη ΓΑΜΑ ΔΕΛΤΑ Εμπορίου και ο κύριος Βατμίτσκη, που είναι υφυπουργός οικονομικών της Ουκρανίας. Ε, Ω προ το γλωσσικό καθεστώ, είναι οι γλώσσε που συνήθω έχουμε στι συνεδριάσει επιτροπή μα, καθώ και τα ουκρανικά. Ε, αναμεταδίδεται ζωντανά στο διαδίκτυο συνήθω η συνεδρίαση. Χωρίς ε, περαιτέρω καθυστέρηση θα ήθελα να ακούσουμε τον Επίτροπο Ντεγκούχτ που έρχεται πλέον τακτικά είναι θαμώνα τη Επιτροπή μα. Καλώ ορίσατε. Σα ακούμε για λίγα λεπτά για την εισαγωγική σα παρουσίαση. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κυρία Μορέρα και πρώτε αντιπρόεδρε κύριε Κλούγεφ, επίσης ε, κύριε Υπουργέ Νταμπρόφσκι, ε, ε, και κυρίες Ευρωβουλευτές πριν 20 χρόνια ε, ε, ε, βρήκε την ελευθερία, ξαναβρήκε την ελευθερία η Ουκρανία πράγμα το οποίο ήταν θετικό και για την Ευρώπη στο σύνολό της πέραν της χώρας Τώρα όμως βρισκόμαστε στο, ε, την παραμονή μιας σημαντικής συμφωνίας, μιας εμπορικής συμφωνίας ορόσημο με την Ευρωπαϊκή Ένωση ε, στα πλαίσια της Συμφωνίας Συνδέσεως, πράγμα το οποίο θα αποτελέσει ένα πρότυπο για τις οικονομικές μεταρρυθμίσεις και θα βοηθήσει να υπάρξουν ε, νέα επίπεδα ε, συνεργασίας εις ε, το εμπόριο και την οικονομική ανάπτυξη. Θα μπορέσει να προσεγγίσει τις οικονομίες μας και να δημιουργήσει νέες ευκαιρίες για την Ουκρανία και τους ενδιαφερομένους Ευρωπαίους σε όλους τους τομείς της οικονομίας. Η συμφωνία δηλαδή αυτή συμβάλλει στην μελλοντική ευημερία της Ουκρανίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει προσφέρει πολλαπλές, ε, ε, ε, πολλαπλές φάσης βοηθείας στους ε, ανατολικούς εταίρους της ε, και έχει στηρίξει την ανάπτυξή τους και αυτό είναι διότι οι δικές μας ε, ανατολικές περιοχές έχουν συμβάλει εις την ανάπτυξη όλης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ένα νέο βήμα είναι η στήριξη αυτή της ε, Ουκρανικής Συμφωνίας ε, Συνδέσεως για το εμπόριο και τα οικονομικά θέματα για να μπορέσει να υπάρξει και μεγαλύτερη πέραν της οικονομικής πολιτική ε, ολοκλήρωση πράγμα το οποίο ε, διοργανώνεται στα πλαίσια της πολιτικής γυπνιάσεως και πρέπει να σας πω ότι εχθές το βράδυ ο κύριος Πλούγεφ και εγώ καταλήξαμε σε μία συμφωνία στα βασικά στοιχεία της ε, ε, τελικής ε, εμπορικής συμφωνίας. Υπάρχουν ακόμη ορισμένα θέματα που πρέπει να ρυθμιστούν αλλά ουσιαστικά είναι έτοιμη η συμφωνία και τώρα εξαρτάται από την Ουκρανική ηγεσία να δημιουργήσει τις πολιτικές προϋποθέσεις κατά τρόπον ώστε να μπορέσει να υλοποιηθεί αυτή η συμφωνία και ελπίζω ότι πολύ σύντομα αυτό θα συμβεί. αυτή η εμπορική συμφωνία θα μας επιτρέψει να ολοκληρώσουμε τη συμφωνία συνδέσεως και ιδίως ε, να ε, ολοκληρώσουμε μέχρι το τέλος του χρόνου την ε, ζώνη ελευθέρου εμπορίου αρκεί να υπάρξουν οι πολιτικές προϋποθέσεις για να μπορέσει αυτό να υλοποιηθεί και στην πράξη περί τίνους ε, διαπραγματευόμαστε ουσιαστικά. Καταρχήν προβλέπουμε το, το άνοιγμα των αγορών για τα εμπορεύματα και τις υπηρεσίες αλλά προχωρούμε και πολύ περαιτέρω Πρέπει να εξετάσουμε ε, τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν πίσω από τα σύνορα για να μπορέσουμε να λύσουμε τα προβλήματα και να αυξήσουμε το, τις εμπορικές συναλλαγές. Η παραδείγματος χάνει τα αγροτικά προϊόντα πρέπει να πληρώνουν δασμούς και ε, να ανταποκρίνονται ε, σε προδιαγραφές. Οι δασμοί μπορούν μπορούν να μειωθούν ή να καταργηθούν αλλά πρέπει να βελτιωθούν και οι προδιαγραφές για το κρέας και το γάλα. Ε, τέτοια προβλήματα θα συζητήσουμε σε θέματα τα οποία αναφέρονται στο εμπόριο. Γι' αυτό και προσπαθούμε να προσεγγίσουμε και να συγκλίνουν οι νομοθεσίες μας επιπλέον θα πρέπει η Ουκρανία να εφαρμόσει τους κανονισμούς ε, και πέραν της καταργήσεως των ε, εισαγωγικών δασμών θα πρέπει να πούμε ότι η Ευρωπαϊκή ε, Ένωση είναι η μεγαλύτερη εμπορική αγορά και η συμφωνία συνδέσεως με την Ουκρανία θα αναφέρεται σε πάρα πολλά θέματα για τις, τους δημόσιους μειοδοτικούς διαγωνισμούς, για τις κυβερνητικές ε, συμβάσεις και ε, θα πρέπει η σχετική νομοθεσία ε, στην Ουκρανία να προβλέπει τα ίδια με αυτή της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και ε, θα πρέπει να ανοίξει η αγορά και στην περίπτωση αυτή η οικονομική ολοκλήρωση και ε, ο εμπορικός στόχος είναι ο πλέον φιλόδοξος που προσπαθεί να επιτύχει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Προσπαθούμε δηλαδή να βελτιώσουμε ε, τις ελεύθερες συναλλαγές με τη χώρα αυτή. Να υπάρχει ένα δια διαφανές ε, ε, περιβάλλον για τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις και στις δύο αγορές. Θα πρέπει ε, να εξυγχρονιστούν το ρυθμιστικό πλαίσιο για να προωθηθούν οι οικονομικές οικονομικές ε, ε, διατάξεις και θα πρέπει ε, να ξέρει ο κάθε ενδιαφερόμενος πότε πρόκειται να υπάρχει μία μεταρρύθμιση και γιατί. Διότι προσπαθούμε να μειώσουμε και τον κίνδυνο για να ανταποκριθούμε στις σύγχρονες επιταγές για τις κεφαλαϊκές επενδύσεις. Γνωρίζετε όλοι ότι οι κεφαλαγορές ε, ε, αυτή την εποχή πιέζονται πάρα πολύ και αυτή η συμφωνία DCFTA προβλέπει ε, διατάξεις οι οποίες θα ανοίξουν την πόρτα της Ουκρανίας στους Ευρωπαίους επενδυτές. Βέβαια πρέπει να σας πω ότι όλα αυτά αναφέρονται στη γενική μας ε, συνεργασία με την Ουκρανία και οι πρόσφατες εξελίξεις στο Κίαβο έχουν θέσει σε κίνδυνο αυτές τις διαπραγματεύσεις αλλά δεν θέλουμε ε, να ε, γυρίσουμε την πλάτη σε αυτή τη χώρα. Θέλουμε να συνεχίσουμε το διάλογο και τα θέματα να συνεχίσουν να συζητούνται. Μόνο όταν θα, έχει, όταν θα υπάρχει μία συμφωνία, ένα σχέδιο συμφωνίας, δηλαδή σαν αυτό που υπάρχει τώρα, θα ξέρουμε πώς και τι μπορεί να χαθεί αν δεν προχωρήσουμε. Προσπαθούμε να ολοκληρέσουμε τη συμφωνία συνδέσεως για την ζώνη ελευθέρου εμπορίου μέχρι το τέλος του χρόνου και μετά θα κάνουμε ένα απολογισμό να δούμε πού βρισκόμαστε. Ε, κυρίες και κύριοι, ο Υπουργός Κλούγεφ και εγώ γνωρίζουμε ότι δεν ε, διαπραγματευόμαστε σε ένα κενό. Είναι ένας δύσκολος, μια δύσκολη εποχή για την οικονομία παντού ε, και υπάρχουν διέξοδα μετά από δέκα χρόνια. Υπάρχουν όλο και περισσότερο προστατευτικά μέτρα παντού. Προσπαθούμε λοιπόν να ε, καταπολεμήσουμε αυτόν τον προστατευσιμισμό και ε, προσφάτως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε την τελευταία έκθεση της εποπτείας των περιοριστικών μέτρων και ε, βλέπουμε ότι το εμπόριο αυξήθηκε κατά 30% με τους ομολόγους Ευρωπαϊκής Ενώσεως αλλά μόνο 17% από τα μέτρα που ξεκίνησαν από την αρχή της κρίσεως έχουν εκπνεύσει. Υπάρχουν όμως πολλά μέλη του G20 που αρχίζουν να χρησιμοποιούν εναλλακτικά μέτρα και αυτό ιδίως σχετικά με τις ε, δημόσιες προμήθειες. Γι' αυτό και θέλουμε ε, να υπενθυμίσουμε εις τους εταίρους ότι έχουν αναλάβει υποχρεώσεις. Πρέπει να βελτιώσουμε λοιπόν τις διμερείς μας σχέσεις για να μπορέσουμε να κρατήσουμε μακριά τις προστατευτικές δυνάμεις και είναι πολύ σημαντικό εφόσον υπάρχουν προκλήσεις οικονομικές η Ευρώπη να μην εφησυχάζει. Εμείς δεν θέλουμε να εφησυχάζουμε με κλειστές αγορές αντιθέτως θέλουμε να είμαστε ανοιχτοί και διαθέσιμοι για το ελεύθερο εμπόριο να ρέει το εμπόριο και να διακινείται και ιδίως λόγω των οικονομικών δυσχεριών χρειαζόμαστε το διεθνές εμπόριο περισσότερο παρά ποτέ για να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε μια επιτυχή έκβαση. Άρα η μέθοδος στην οποία σκεπτόμαστε εις ε, τα πλαίσια αυτής της συμφωνίας θα είναι επικερδής και για την Ουκρανία και για εμάς θα βελτιώσει την ε, Ουκρανική οικονομία και θα αποτελέσει ένα ορόσημο διότι θα επιβεβαιώσει τις κοινέ μας αξίες και ελπίζουμε ότι τις επόμενες εβδομάδες και μήνες θα μπορέσουμε να υλοποιήσουμε αυτή τη συμφωνία. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Δεν θα μπορούσαν να ήταν καλύτερα τα πράγματα. Δηλαδή, μας είπατε ότι οι διαπραγματεύσεις για τη σύναψη εμπορικής συμφωνίας, συμφωνίας ελευθέρων συναλλαγών έχουν προχωρήσει και αυτό είναι πολύ καλό νέο. Και το γεγονός ότι προωθήθηκε το θέμα αυτό είναι η καλύτερη μαρτυρία για την πολιτική μας ελευθέρων συναλλαγών. και χαιρόμαστε που κάνατε αυτή την ανακοίνωση εδώ και τώρα. Τώρα ας ακούσουμε τον κύριο Κλούγεφ, ο οποίος είναι Υπουργός Οικονομικής Ανάπτυξης και Εμπορίου, πρώτος αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και με χαρά θα ακούσουμε την άποψή σας, τις απόψεις σας για τα συμπεράσματα της συμφωνίας, για τη σύναψη της συμφωνίας. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Μορέιρα, κύριε Επίτροπε, κύριε Ντεγκούχτ, κυρίες και κύριοι, Είμαι ευγνώμων στους διοργανωτές γιατί μας δίνεται την ευκαιρία να μιλήσουμε για θέματα ύψης της εμπορικής σημασίας μέσα στα πλαίσια της διαδικασίας ολοκλήρωσης των διαπραγματεύσεων για τη δημιουργία μίας εις βάθος και συνεκτικής συμφωνίας ελευθέρων εμπορικών συναλλαγών. Είχαμε αρχίσει τις διαπραγματεύσεις το 1997 και θα ήθελα να σας επιβεβαιώσω ότι χτες το βράδυ μετά από εντατικές διαπραγματεύσεις μπορέσαμε να κλείσουμε τη συμφωνία ως προς τα βασικά σκέλη της, δηλαδή την συμφωνία αυτή ελευθέρων συναλλαγών. Οι συμφωνίες και η συμφωνία με τον Επίτροπο Ντεγκούχτ θα οδηγήσουν σε θετική έκβαση μέχρι το τέλος του έτους. Και νομίζω ότι πρόκειται για μια συμβολική σημασίας συμφωνία. Είπαμε στους εμπειρογνώμονες ότι θα πρέπει να ε, προσπαθήσουν να φτάσουν σε αίσιο πέρα ως προς την συμφωνία αυτή. Και σας ευχαριστώ πολύ για τις προσπάθειές σας. Τώρα, σε σχέση με τις διαπραγματεύσεις αυτές που διήρκεσαν τριάμιση χρόνια, δείχνουν ότι υπάρχουν δυνατότητες οι οποίες σχετίζονται με όλα τα σκέλη της συμφωνίας και της εφαρμογής σας. Και αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς, έτσι ώστε να φτάσουμε στην ε, οικονομική ολοκλήρωση μέσω της ε, εμπορικής αυτής ε, συμφωνίας για την ευημερία των ε, πολιτών της Ουκρανίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν θα πρέπει όμως να αρνηθώ ότι οι διαπραγματεύσεις ήταν ιδιαίτερα δύσκολες και ευτυχώς φτάσαμε σε συνένεση σε όλα τα θέματα ως προς τις υπηρεσίες, τα αγαθά, τις συναλλαγές στον ενεργειακό τομέα, την αμοιβαία προστασία του εμπορίου, του ενεργειακού τομέα, του τομέα του ανταγωνισμού, των κρατικών ενισχύσεων και μιλήσαμε, μάλλον ε, και συμφωνία ως προς τις δημόσιες προμήθειες καθώς και ε, δασμολογικού χαρακτήρα συμφωνία. Γνωρίζουμε ότι θα υπάρξει μία μεταβατική περίοδος σε σχέση με τις συναλλαγές στο εμπόριο, στα αγαθά, στις υπηρεσίες, όπου θα πρέπει να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στο κοινοτικό και εκτιμένο. Και βεβαίως πάντα θα πρέπει κανείς να φτάσει σε συμβιβασμούς, διότι στην ιστορία της διπλωματίας πάντα βλέπουμε ότι μόνο μέσω συμβιβασμών επιτυγχάνεται κάτι. Στην περίπτωση των δικών μας διαπραγματεύσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση είμαι πολύ ευτυχής για αυτό τον συμβιβασμό και θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Επίτροπο Ντεγκούχτ για την προσωπική του συνεισφορά για αυτή την επιτυχία. Το συνολικό ο, ισολογισμός και μάλλον το ισοζύγιο, θα μπορούσα να πω αυτή τη συναλλαγή, είναι θετικό και για τη μία πλευρά και για την άλλη. Η Ουκρανία θα ήθελε να έχει πρόσβαση στην ευρωπαϊκή αγορά με 500 εκατομμύρια καταναλωτές και εσείς φυσικά θέλετε να μπορέσετε να εισδύσετε στη δική μας αγορά γιατί διαθέτουμε πολλούς πόρους και ξέρετε ότι οι συναλλαγές σας με την Ουκρανία ανέρχονται στο 30% των συνολικών συναλλαγών. Αυτό που έχει σημασία είναι να αρθούν οι δυσχέρειες των Ουκρανών εξαγωγέων στην Ευρωπαϊκή Αγορά και τούμπαλιν. Όπως ελέγχθη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εμείς ζητήσαμε τη μεγαλύτερη δυνατή απελευθέρωση για την αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πρόσβαση χωρίς προσκόμματα στη δική μας αγορά. Αυτό που έχει σημασία λοιπόν είναι και οι εισαγωγές τεχνολογιών εχμής για να απτύξουμε τη βιομηχανία μας και την συνεχή ανάπτυξη της οικονομίας μας. Αντιμετωπίζουμε βασικά καθήκοντα και ε, βασικά ζητήματα αρμοδιατήτων μέσα στα πλαίσια, σε αυτής, ε, μέσα στα πλαίσια αυτής της συμφωνίας. Και θα πρέπει να εναρμονίσουμε την ε, νομοθεσία μας και να προβούμε και σε συστημικού χαρακτήρα μεταρρυθμίσεις. Αυτό ακριβώς προσπαθούμε να επιτύχουμε σε κάθε τομέα της οικονομίας μας. και μέσω αυτής της Συμφωνίας Ελευθέρων Συναλλαγών θα προωθήσουμε συγκεκριμένα σχέδια για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε και νομοθετικά. Θα ήθελα να σας πω για τα μέτρα που λαμβάνουμε για τις ελεύθερες συναλλαγές με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Προσπαθήσαμε το καλοκαίρι να προβούμε σε μεταρρυθμίσεις έτσι ώστε να υπάρχουν ευεργετήματα στα πλαίσια αυτής της σφαιρικής και σε βάθος συμφωνίας ελευθέρων συναλλογών. Αυτό αφορά τη διατροφική ασφάλεια, την ποιότητα τροφίμων, ε, τα οποία τρόφιμα αυτά θα πρέπει να ανταποκρίνεται στα ε, πρότυπα και τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, θα πρέπει να υπάρχει και ανταπόκριση στα δεδομένα και στις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς τα ενεργειακά προϊόντα. Μιλήσαμε για μια συμφωνία ελευθέρων συναλλαγών όπου υπησέρχονται όχι μόνο οικονομικοί παράγοντες, αλλά και παράγοντες πολιτικού χαρακτήρα. Αυτό που έχει σημασία λοιπόν είναι ότι θα πρέπει να φτάσουμε και σε υψηλές προδιαγραφές δημοκρατίας, οικονομικό ανταγωνισμό και να τηρούνται και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η Ουκρανία και η Ευρώπη έχουν μια κοινή ιστορία και αξίες. Μέσα στα πλαίσια αυτής της ε, σφαιρικής και σε βάθος συμφωνίας ελευθέρων συναλλαγών θα κάνουμε το πρώτο βήμα έτσι ώστε να συσπηρωθούμε, να προσεγγίσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση και σας ευχαριστούμε για τη βοήθειά σας. Ευχαριστούμε πολύ, λέει ο κύριος θα θέλαμε να ακούσουμε τώρα ε, τον εκπρόσωπο της Πολωνικής Προεδρίας ε, του Συμβουλίου, διότι έχουν επενδέσει πολλά από πολιτικής πλευράς για την ενίσχυση της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και θα πρέπει να μοιραστούμε την επιτυχία. Συγχαρητήρια. Κύριε Κόρολετς, είστε η Υφυπουργός Οικονομικών Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Πιστεύω ότι τα εύσημα θα πρέπει να αποδοθούν ε, κατά κύριο λόγο στους διαπραγματευτές ε, του τέστην, στον Επίτροπο Ντεγκού. Σε χαρητήρια και στον ε, κύριο Κλούγεφ, τον Υπουργό παρά τον Πρωθυπουργό. Θα ήθελα να δηλώσω ικανοποιημένος με την έκβαση των, και το πέρας των διαπραγματεύσεων. Ε, χαιρόμαστε με αυτά τα καλά νέα. Ε, πιστεύω ότι με τα γεγονότα των τελευταίων ημερών όλοι θα εξετάσουμε υπό νέο φως ε, τις ε, διαπραγματεύσεις. Θα πρέπει να συνεργαστούμε, όπως σωστά είπατε, για να ε, δημιουργήσουμε πρόσφορες σε πολιτικές συνθήκες που θα μας επιτρέψουν να υιοθετήσουμε αυτή τη συμφωνία. Κατά τη γνώμη μας, η ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων για τη σύναψη αυτής της ε, συμφωνίας DCFTA, καθώς και ε, ε, η διοργάνωση της Συνόδου το Δεκέμβριο φέτος στο Κίεβο θα μας βοηθήσουν να υλοποιήσουμε τους στόχους της ανατολικής εταιρικής σχέσης. Η Πολωνική Προεδρία θα ήθελε να διασφαλίσει σταθερότητα στην περιοχή ως προς την νότια και την ανατολική διάσταση αυτής της εταιρικής σχέσης. Όπως ακούσαμε, το κλειδί και ο πλέον αποτελεσματικός τρόπος για την ενίσχυση των εμπορικών σχέσεων είναι η ολοκλήρωση. Ολοκλήρωση μέσα από τη συμφωνία DCFTA, δηλαδή η βάθος και σφαιρική συμφωνία ελευθέρων εμπορικών συναλλαγών, με τη σταδιακή κατάργηση των εμπορικών φραγμών, ε, αλλά όχι μόνο μέσω από ρυθμιστικές προσαρμογές σε τομείς όπως ε, οι κρατικές προμήθειες, ε, οι τελωνιακές διασαφήσεις και διαδικασίες, ε, πολιτική ανταγωνισμού, ε, διαγωνισμοί. Θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας ε, στο ότι η Ουκρανία είναι η χώρα που έχει ε, σημειώσει τα μεγαλύτερα επιτεύγματα στη διαδικασία ολοκλήρωσης. Αν εξετάσουμε δηλαδή τις υπόλοιπες χώρες που μετέχουν σε αυτήν την ανατολική εταιρική σχέση θα διαπιστώσουμε ότι η Ουκρανία έχει κάνει σοβαρά βήματα προς μια γενικότερη οικονομική ολοκλήρωση. Αυτό αποδεικνύεται από την προσχώρησή της στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου εμπορίου ήδη από το 2008. Η Ουκρανία επίσης ε, σταδιακά προσαρμόζει και το ένομο σύστημά της ε, στους ευρωπαϊκούς ε, κανόνες και πρότυπα. Επ' αυτού θα μπορούσα να σας δώσω παραδείγματα όπως η συνεργασία και η υιοθέτηση προτύπων και κανόνων Ε, ως προς ε, την αμοιβαία δικαστική αρρωγή, συνδρομή παραδείγματος χάρη ή την συνεργασία στα φορολογικά ζητήματα, στην υιοθέτηση των κατευθυντηρίων γραμμών ε, του ΠΟΕ σε σχέση με τις πολυεθνικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην επικράτειά της. Επίσης, συνειδητοποιούμε ότι οι αρμόδιες αρχές θέλουν να αρχίσουν να εργάζονται για να υιοθετηθεί η σύμβαση όσα ε, για την καταπολέμηση ε, της ε, διαφθοράς στους ανώτερους, σε επίπεδο ανώτερων αξιωματούχων και ονομάζεται αυτό Σύμβαση κατά της δωροδοκίας. Έτσι την έχουν ονομάσει. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που ασθενίζονται το πνεύμα των εργασιών του ΟΣΑ στην Ουκρανία και ευελπιστούμε ότι θα ενισχυθεί αυτή η συνεργασία. Ε, και η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ουκρανία θα επωφεληθούν ε, από την σύναψη της ε, συμφωνίας DCFTA με την υιοθέτηση αυτής της εμπορικής συμφωνίας σταδιακά θα ενταχθεί η Ουκρανία ε, στην ευρωπαϊκή αγορά με την κατάργηση ε, των φραγμών ε, ως προς τα αγαθά και τις υπηρεσίες και θα διευκολυνθεί η διακίνηση των κεφαλαίων. Αυτό είναι υποφελές για τους επενδυτές και τους επιχειρηματίες αμφωτέρων των πλευρών διότι θα δημιουργηθούν βίωνες συνθήκες για τις επιχειρήσεις. Οι καταναλωτές επίσης θα είναι κερδισμένοι διότι θα έχουν πρόσβαση σε ασφαλέστερα προϊόντα. θα έχουμε επίσης ε, ένα καλύτερο επίπεδο προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων. Με την υπογραφή της ε, συμφωνίας DCFTA, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα εξασφαλίσει πρόσβαση σε μία αγορά σχεδόν 50 εκατομμυρίων καταναλωτών, καθώς ε, και ευκαιρίες για να υλοποιήσει επενδυτικά σχέδια σε μια οικονομία με αναπτυξιακό ρυθμό έως και 5% για το τρέχον έτος. Ε, ο συνδυασμός ε, της δυναμικής αυτής ανάπτυξης σε συνδυασμό με το μέγεθος της ε, Ουκρανικής οικονομίας ε, δύναται να παράσχει στην ευρωπαϊκή οικονομία σημαντικότατα ωφέλη και αναπτυξιακό δυναμικό. Αφετέρου, η ουκρανική οικονομία, πέρα από την απελευθέρωση της πρόσβασης ε, στην αγορά της Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης, μέσω της υιοθέτηση διαφανών κανόνων για τη λειτουργία των επιχειρήσεων, μπορεί κάλλιστα να προσελκύσει μεγαλύτερο αριθμό αλλοδαπών επενδύσεων, ε, κυρίως ε, όσον αφορά σε επενδύσεις ε, στην υποδομή. Οι επιχειρήσεις θα προσαρμοστούν, οι αγορές θα προσαρμοστούν, η υιοθέτηση όλων αυτών των κανόνων θα γίνει με σταδιακό τρόπο, είναι προφανές. σχετικά με την εφαρμογή των κανόνων του ΩΣΑ στην Ουκρανία κυρίως. Ε, το επόμενο βήμα Μόλις δηλαδή υπερατωθούν οι διαπραγματεύσεις για τη σύναψη της DCFTA και με στόχο να ενισχύσουμε την οικονομική συνεργασία και τη βελτίωση του επιχειρηματικού κλίματος, το επόμενο βήμα λοιπόν θα έπρεπε να είναι η υπογραφή ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ουκρανία μια συμφωνία για την προστασία αυτών των επενδύσεων. Ε, αν κρίνουμε από την εμπειρία της ε, Πολωνίας ε, τα τελευταία 12 χρόνια θα μπορούσε ε, κάποιος να καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η εσωτερική αγορά είναι καλύτερη κινητήριο αναπτυξιακή δύναμη και το καλύτερο εχέγγυο για την ασφάλεια και την σταθερότητα για όλους τους οικονομικούς φορείς. Οπότε η οικονομική ολοκλήρωση της Ουκρανίας είναι προς όφελος και της Ένωσης και της Ουκρανίας. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε πολύ. Άρα έληξε η παρουσίαση των θεμάτων μας με βάση, τους, ε, με βάση αυτά που μας είπαν οι προσκεκλημένοι μας. Έχουμε πέντε λεπτά γιατί σε λίγα λεπτά ο κύριος Δεκούχ πρέπει να αποχωρήσει. Το γνωρίζαμε εξ αρχής. Θα μπορέσουν να υποβληθούν ερωτήσεις από την Επιτροπή Ίντα προς τους προσκεκλημένους μας. Ας αρχίσουμε με ερωτήσεις προς τον Επίτροπο, με τηλεγραφικές ερωτήσεις και ε, λόγο έχει ο κύριος Ζαλεύσκη, ο Παύλ Ζαλεύσκη, ο οποίος είναι εισηγητής της Επιτροπής μας για τις συστάσεις αυτές. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Θέλω καταρχήν να συγχαρώ τον κύριο Ντεγκούχ και τον κύριο Κλούγεφ και θέλω να ευχαριστήσω τον πρόεδρο που οργάνωσε αυτή την εκδήλωση και, για την προσωπική του συμβολή σε αυτή. Ε, έχω να θέλω να αναφερθώ στις εμπορικές σχέσεις, δηλαδή ε, στην ε, υπογραφή της συμφωνίας μεταξύ Ευρωπαϊκής Ενώσεως και Ουκρανίας η οποία θα ολοκληρωθεί σύντομα ελπίζω και μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας η οποία έχει ήδη υπογραφεί την τρίτη μάλιστα για να είμαι συγκεκριμένος θα ήθελα να ρωτήσω πώς αυτές οι δύο συμφωνίες οι οποίες θα υλοποιηθούν σύντομα πώς θα ε, έχουν επιπτώσεις στις ε, αμοιβέ εμπορικές σχέσεις και στην οικονομία της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Κάποιο άλλο μέρος της Επιτροπής ο κύριος Κούτας και ο κύριος Σόλτς από την ΓΟΕ. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, και κύριε Επίτροπε ε, έχουμε όντως ε, ένα πολύ προκλητικό πρόγραμμα για να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε αυτή την ε, Συμφωνία Ελευθέρου Εμπορίου. Ε, ποια είναι η σχέση μεταξύ του FTA και ε, της συμφωνίας συνδέσεως. Ε, έχετε αντιληφθεί ότι πρέπει να υπάρξει κοινή συνεννόηση αλλά πέραν αυτού να προχωρήσει η οικονομική και εμπορική συμφωνία. Δηλαδή θα ήθελα να ξέρω πού βρισκόμαστε στο θέμα αυτό. Και επίσης πρέπει να καλύψουμε και άλλα θέματα. Ξέρω ότι ο χρόνος είναι περιορισμένος. Μπορείτε λοιπόν να μας δώσετε ένα παράδειγμα για το πώς θα καλύψετε την συμφωνία στο γεωργικό τομέα. Ο κύριος Κλούγεφ μπορεί να μείνει περισσότερα, οπότε μπορούμε να συνεχίσουμε με τις ερωτήσεις προς αυτόν αφού φύγει ο, ο Επίτροπος Ντεγκούφ, το οποίο έχει ακόμη λίγα λεπτά, κανένα δεκάλεπτο, όχι παραπάνω. Ο κύριος Πάβελ Κόβαλ ο οποίος είναι ο επικεφαλής της ε, ε, κοινοβουλευτικής ε, αντιπροσωπείας της Ουκρανίας. Και εγώ έχω μία ερώτηση σχετική με αυτή που μόλις ετέθηκε, δηλαδή να μας δοθούν συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με τα εμπόδια που υπάρχουν ακόμη από πλευρά Ουκρανίας και Ευρωπαϊκής Ενώσεως για να ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις και να ακυρωθεί η συμφωνία. Άλλο μέλος της Επιτροπής Ίντα, αν όχι, θα δώσω το λόγο στον κύριο Άντριαν Σεμπάσιαν, ο οποίος είναι επίσης Ευρωβουλευτής. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ για την παρουσίασή σας κύριε Επίτροπε. Ήταν εξαιρετική. Είπατε ότι δεν εργάζεστε στο κενό. Αναφέρατε την κρίση. Αλλά αναρωτιέμαι μήπως θα έπρεπε επίσης να έχουμε υπόψη μας τον ανταγωνισμό. Και εδώ αναφέρομαι στον, στον ανταγωνισμό μεταξύ της προσφοράς της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και της προσφοράς για να είμαι σαφής της Ρωσίας για μία συμφωνία εμπορική και μήπως γι' αυτό δεν θα έπρεπε να επιταχύνουμε ε, την ολοκλήρωση της δικής μας συμφωνίας για να παραμείνει η Ουκρανία με το μέρος μας. Επίσης ε, αντιλαμβάνουμε ότι όταν οι συνθήκες θα το επιτρέψουν θα ολοκληρωθεί η συμφωνία αλλά ε, ε, δεν θεωρείται ότι υπό τις ε, συνθήκες που διέπουν την οικονομία είναι υποχρεωτικό να καταλήξουμε σε αυτή τη συμφωνία και το, η συμφωνία αυτή να αποτελέσει ένα, πρόβλη, ένα πρότυπο για να μπορέσουν ορισμένες χώρες να συμμορφωθούν με τις αρχές μας. Ευχαριστώ. Κύριε Επίτροπε, σας ευχαριστώ και χαίρομαι που μπορείτε να μείνετε λίγα λεπτά παραπάνω για να απαντήσετε σε αυτές τις ερωτήσεις. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι. Ε, η κοινοπολιτεία ανεξαρτήτων κρατών συμπεριλαμβανομένη και τη Ουκρανία φυσικά έχουν τη δυνατότητα να συνάπτουν τέτοιε εμπορικέ συμφωνίε σε δυνάμει και των οικονομικών προτεραιότητων προτεραιοτήτων τους ε, και ε, θα συνάψουμε αυτή τη συμφωνία με την Ουκρανία, αλλά όχι μόνο. Στο παρελθόν έχουν υπάρξει τέτοιες συμφωνίες και το ίδιο προβλέπεται και για το μέλλον. Είναι ανεξάρτητη η χώρα η Ουκρανία και θα αποφασίσει φυσικά μόνη της τι είδους συμφωνίες θέλει να συνάψει. Να σημειώσουμε παρεπιπτόντω ότι όλες αυτές οι χώρες της κοινοπολιτεία ε, ανεξαρτήτων ε, κρατών ε, έχουν τέτοιου είδου συμφωνίες με την πρώην Σοβιετική Ένωση και τώρα επικαιροποιούνται σταδιακά όλε αυτές οι παρελθούσε συμφωνίες. Η Ρωσία έχει υπογράψει συμφωνία με άλλες 7 πρώην Σοβιετικές Δημοκρατίες για την κατάργηση εισαγωγικών και εξαγωγικών δασμών για μια σειρά προϊόντων. Ανακοινώθηκε δε η συμφωνία μετά από ε, τις συνομιλίες στην Αγία Πετρούπολη ε, και ε, το Καζακστάν, η Αρμενία, το Κυργιζιστάν, η Μολδαβία και το Τατζικιστάν μεταξύ αυτών των χωρών δεν έχουμε λεπτομέρειες για το περιεχόμενο αυτών των συμφωνιών. Δεν ξέρουμε ακριβώς ε, δηλαδή ποια προϊόντα θα καλυφθούν, αλλά ε, υπό φυσιολογικές συνθήκες πρόκειται μόνο για αγαθά και αυτό ε, συνιστά και τη βασικότερη διαφορά με τη δική μας συμφωνία που είναι σφαιρική και εις βάθος. Μέχρι το τέλος του 2011 το Ουσβεγιστάν, το Τουρκμενιστάν και το Αζερβαϊτζάν ενδέχεται να προσχωρήσουν σε αυτή τη συμφωνία. Αυτή η Συμφωνία Ελευθέρων Εμπορικών Συναλλαγών θα πρέπει να κυρωθεί από το Κοινοβούλιο των χωρών που μέχρι στιγμή έχουν υπογράψει αυτή τη συμφωνία. Ε, προτού τεθεί σε ισχύ το 2012. Έτσι έχουν τα πράγματα και δεν διαβλέπω καμία δυσκολία. Ε, είμαι αισιόδοξο ε, και θεωρώ ότι η συμφωνία DCFTA θα είναι πραγματικά σφαιρικότερη και πιο εις σε σχέση με τις συμφωνίες με της πρώην Σοβιετικής Δημοκρατίας ε, που έχουν υπογραφεί με τη Ρωσία. Η DCFTA, αυτή η συμφωνία, εντάσσεται στην Συμφωνία Σύνδεσης Ευρωπαϊκής Ένωσης Ουκρανίας, η οποία θα πρέπει να οριστικοποιηθεί προτού ε, προς υπογραφή η DCFTA. Ε, είναι η συνήθις ε, πρακτική και δεν υπάρχει κανένας ε, λόγος, δεν συντρέχει λόγος για να τροποποιήσουμε αυτή τη διαδικασία. Η συμφωνία σύνδεσης, οι διαπραγματεύσεις μάλλον για τη συμφωνία σύνδεσης είναι υπό την αρμοδιότητα της Βαρόνης Άστον, αλλά προφανώς η DCFTA είναι βασικό δομικό κομμάτι της ε, συμφωνίας ε, σύνδεσης, ε, δηλαδή η DCFTA, αν θέλετε, είναι το κτίριο και η Συμφωνία Σύνδεσης η στέγη. νομίζω ότι αυτή η εικόνα μπορεί να σας μεταφέρει καλύτερα το, το μήνυμα. Θα προσπαθήσουμε να ολοκληρώσουμε τη Συμφωνία Σύνδεσης μέχρι το τέλος του 2011 επίση, αλλά όπως ε, προείπα η DCFTA και η Συμφωνία Σύνδεσης ε, δεν ε, τελούν αντικείμενο διαπραγματεύσεων σε κενό αέρος αν θέλετε, αλλά λειτουργούμε μέσα σε ένα δεδομένο πολιτικό πλαίσιο και όπως σαφέστατα ξεκαθάρισα στα εισαγωγικά μου σχόλια έχουμε πλέον ένα κείμενο για την DCFTA, έχουμε όλε τι λεπτομέρειε. Έχουν δηλαδή ολοκληρωθεί, αν θέλετε, οι διαπραγματεύσει, αλλά για να ε, πάρει σάρκα και οστά αυτή η συμφωνία, η Ουκρανία ε, θα χρειαστεί να δημιουργήσει τις ε, κατάλληλες πολιτικές συνθήκες. Αν μπορέσουμε εμείς να συνδράμουμε την Ουκρανία δεν θα αντιστάσουμε, αλλά ε, δεν μπορούμε παρά να αναγνωρίσουμε ότι υπάρχει ένα σοβαρότατο πρόσκομα αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, ε, ο, οι πολιτικοί ηθήνοντες ε, της Ουκρανίας θα πρέπει να κάνουν τα δέοντα και σας είπα ο κύριος Φαν ο κύριος Μπαρόσο και η Βαρόνη Άστον από ευρωπαϊκής πλευράς έχουν την πλήρη αρμοδιότητα για αυτή την συμφωνία. Υπάρχει αυτός ο ανταγωνισμός με τη Ρωσία, στον οποίο αναφέρθηκαν οι συνάδελφοι. Πρώτον, αυτό που χρειαζόμαστε είναι μια καλή συμφωνία. Νομίζω ότι είναι και το πρωταρχικό μας μέλημα. Ε, προφανέστατα δεν υπάρχει προηγούμενο. Εδώ και 7 χρόνια επεξεργαζόμαστε αυτή τη συμφωνία. Οδηγεί σε σύγκληση ε, νομοθεσία. Είναι πολύ λεπτομερή συμφωνία. Είναι ει είναι σφαιρική. Πρόκειται για συμφωνία νέα γενιά, θα την αποκαλέσω έτσι. Δεν θεωρούμε ότι υπάρχει λοιπόν ανταγωνισμός. Ε, αντίθετα, είμαστε στα πλαίσια μιας ευρείας διαδικασίας ε, που θα οδηγήσει σε μεγαλύτερη ολοκλήρωση των ευρωπαϊκών κρατών και σε μια ευρεία διαδικασία ε, σε ολοκλήρωση, ούτω ώστε η ανατολική εταιρική σχέση να ενταχθεί στον ευρωπαϊκό χώρο. Αυτό επιδιώκουμε και ξαναείπα ότι είναι βασικό δομικό στοιχείο αυτή η συμφωνία ε, DCFTA στο συνολικό οικοδόμημα. Ε, υπό αυτή την οπτική γωνία θα πρέπει να εξεταστεί η συμφωνία. Ω προ τη Γεωργία, έχουμε πολλούς επιμέρους τομείς. Φυσικά η πολύ σημαντική νομοθεσία για τα, τα πρότυπα, SPS. Ε, που ισχύει και, μπορεί, και επιτρέπει συγγνώμη, ε, τις εμπορικές συναλλαγές ε, για τα τρόφιμα και για τα γεωργικά προϊόντα. Επίσης, καλύπτονται και άλλα προϊόντα όπου θα κλείψουν εισαγωγικοί δασμοί, τα TRQs παραδείγματος χάρη, έτσι ονομάζονται. Πρόκειται για συγκεκριμένες δασμολογικές ποσοστώσεις, δηλαδή μπορεί κάποιος να εξάγει και να εισάγει ε, τηρώντας μια ποσόσταση ανά κατηγορία ε, προϊόντων ε, με ε, προτιμησιακούς δασμούς. Δεν νομίζω ότι έχει νόημα τώρα να επισέλθω σε λεπτομέρειες για τις τεχνικές διατάξεις της συμφωνίας. Ε, προφανέστατα είναι διαθέσιμες όλες οι πληροφορίες για τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με το που ολοκληρωθεί η διαδικασία. Σε ε, πρώτο στάδιο θα πάρει τις πληροφορίες ο εισηγητής σας ε, και κατόπιν ε, θα ακολουθήσει πιο λεπτομερή συζήτηση, αλλά δεν νομίζω ότι είναι το αντικείμενο της σημερινής μας συνάντησης, όλες αυτές τις τεχνικές λεπτομέρειες. Πρόεδρος. Πριν δώσω το λόγο στον κύριο Κλίγεφ, θα ήθελα να αποχαιρετήσω τον Επίτροπο Ντεγκούχτ ε, να προσθέσω επίσης ότι έχουμε την αίσθηση πως είμαστε στην πρώτη εμπορική γραμμή, στο, στο στο πρώτο εμπορικό μέτωπο με αυτή τη συμφωνία. Αντίο. Я хотел бы э, подтвердить э, все, что касается... Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να σας πω ότι θα αναφερθώ στη συμφωνία που υπεγράφει ε, για τις ε, χώρες ε, του CIS επί του οποίου υπάρχουν εδώ και ε, χρόνια ε, διμερείς συμφωνίες πρόκειται για την Ρωσία και τη Μολδαβία την Λευκορωσία και το Καζακστάν και ε, διάφορες άλλες σχετικά με αυτή την ε, κοινοπολιτεία των ανεξαρτήτων κρατών. Προσπαθούμε λοιπόν να ενσωματώσουμε όλες αυτές τις συμφωνίες σε μία γενικότερη συνθήκη και να την υπογράψουμε. Ε, δεν βλέπω λοιπόν πού θα επέμβει ε, το, ε, το η ε, συνθήκη αυτή ε, με την κοινοπολιτεία, με αυτή την εμπορική συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ενώσεως και Ουκρανίας. Θα προσπαθήσουμε να ε, απελευθερώσουμε τα την διακίνηση αγαθών παραδείγματος χάρη να αναφερόμαστε εις ε, τις, ε, στις εξαγωγές δημητριακών κρέατος γεωργικών προϊόντων της ε, Ουκρανίας για το κρασί για το ηλιέλεο και διάφορα άλλα κεφάλαια τα οποία συζητούμε εδώ και πολύ καιρό, πολύ σοβαρά και η συζήτηση αυτή για την ε, γεωργία έχει ξεκινήσει εδώ και πολλά χρόνια αλλά καταλήξαμε ε, πριν από τρεις μήνες. Όλα αυτά έχουν σχέση και με την συμφωνία συνδέσεως και τον ε, ε, χώρο ελευθέρου εμπορίου όπως είπε ο κύριος Ντεγκούχτ. Υπάρχουν λοιπόν διάφορες παράμετροι στην ε, συμφωνία αυτή ε, αλλά πρέπει να πούμε ότι αυτή η συμφωνία είναι μέρος του συνόλου και γι' αυτό καθήκον των Ουκρανών είναι να μπορέσουν να καταλήξουν σχετικά με αυτή τη συμφωνία μέχρι μέχρι το τέλος του χρόνου ε, διότι όπως σας είπα ε, υπάρχει μία συμφωνία επί της αρχής και τώρα θα πρέπει οι δικοί μας να προβούν στην ε, εκπόνευση των λεπτομεριών. Και τώρα ο κύριος Κόβαλτσεκ ο κύριος Κόλοτσεκ μπορεί να απαντήσει στις ερωτήσεις των Ευρωβουλευτών. Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα να σας αναφέρω ότι ότι αν υπάρχει η πιθανότητα σύναψης σφαιρικής και σε βάθος συμφωνίας ελευθέρων συναλλαγών ε, μεταξύ Ουκρανίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και προβάλλουμε νέες ε, απελευθερώσεις συναλλαγών με νέους ε, εμπορικούς και οικονομικούς εταίρους Έχω την εντύπωση ότι αυτό θα ήταν προς μεγάλο όφελος όλων των φορέων, δηλαδή να υπάρχει πρόσβαση στο ελεύθερο εμπόριο. Αυτό είναι ένα από τα βασικά αξιώματα του ελευθέρου εμπορίου. Έτσι διανοίγουμε νέες, νέους ορίζοντες στις οικονομικές δυνατότητες και συναλλαγές και στην οικονομική διπλωματία. Σας ευχαριστώ. Έχουμε λίγα λεπτά στη διάθεσή μας. Πριν αρχίσουμε με το δεύτερο, πριν συνεχίσουμε μάλλον με το δεύτερο τμήμα του σεμιναρίου και ίσως υπάρχουν περαιτέρω ερωτήσεις. Ιδιαίτερα προς τον κύριο Κλούγεφ. Υπάρχουν ερωτήσεις. Φαίνεται πως... Όχι, όχι, υπάρχουν ερωτήσεις. Έχετε το λόγο. Ο κύριος Κόβαλα. Θα ήθελα να δούμε λίγο εις βάθος τα πράγματα. Οι ευρωβουλευτές μπορεί να υποβάλουν πιο λεπτομερείς ερωτήσεις. Υπάρχουν μεγάλα προσκόμματα ως προς τις συζητήσεις μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης Ουκρανίας για τη Συμφωνία Σύνδεσης ο Πάβελ Ζαλεύς και κάτι λέει, αλλά δεν τον ακούω. Θα ήθελα ε, ε, να μου πείτε λοιπόν ότι κατά πόσο υπάρχουν προσκόμματα ναι ή όχι στη Συμφωνία Σύνδεσης. Και σας παρακαλώ να επικρατήσει λίγη ησυχία. Helmut Scholz. Ο Helmut Scholz. Ευχαριστώ. Θα μιλήσω γερμανικά. Έχω ακόμη μία ερώτηση διότι ο Πρωθυπουργό ε, έχει απευθυνθεί και στην Πολωνική Προεδρία για τα θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Ε, τι θα γίνει τώρα με την ε, συμφωνία αυτή. Θα προσχωρήσει η Ουκρανία και στη συμφωνία ΑΚΤΑ σχετικά με την πνευματική πραγματική διεκτησία και την ε, ε, προστασία της αναφέρονται αυτά στα κείμενα της συμφωνίας και σχετικά ε, με την Ρωσία ή άλλους εμπορικούς εταίρους της Ουκρανίας θα θίξει η Ουκρανία τα θέματα αυτά προς τους άλλους εταίρους της γιατί αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία για τη μελλοντική συνεργασία Ευρωπαϊκή Ευρωπαϊκής Ενώσεως και Ουκρανίας. Και πάλι. Εντάχει και πάλι. Γιατί δεν θα ήθελα να παίζονται παιχνίδια. Ξέρουμε όλοι ποια είναι τα προσκόμματα. Αλλά το βασικό ζήτημα είναι πώς θα υπερβούμε αυτά τα προσκόμματα θα το κάνετε δίνοντας μαθήματα από τα υψίπεδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ζητώντας πράγματα που θέλουμε ή θα πρέπει να προτείνουμε ένα σύστημα συνεργασίας. Και εδώ δεν μιλώ για, το εμπόριο, αλλά στη συνεργασία στον τομέα της δικαιοσύνης. Αυτό είναι το ζήτημά μας. Ξέρουμε όλοι ποιο είναι το πρόβλημα. Κάνοντας λοιπόν αυτό το σύνδεσμο μεταξύ εμπορίου και ορισμένων υποθέσεων με συγκεκριμένες κωδικοποιήσεις δεν προχωράμε σωστά και ίσως χάσουμε την ευκαιρία να δούμε την πτυχή του ανταγωνισμού. Με συγχωρείτε για αυτή την παρέμβαση, αλλά γνωρίζουμε όλοι πολύ καλά ε, που είναι τα προσκόμματα και ας μην το παίζουμε ναρκισιστικά. Ο κύριος Κλούγεφ έχει το λόγο για να απαντήσει στο δεύτερο αυτό γύρο ερωτήσεων. Ευχαριστώ για τις ενδιαφέρουσες ερωτήσεις που υποβάλατε. Όσο αφορά, όσον αφορά αυτά τα προσκόμματα τα οποία εξακολουθούν και υπάρχουν σε σχέση με τις ε, συμφωνίες ελευθέρων συναλλαγών υπάρχουν πολιτικά ζητήματα τα οποία θα πρέπει να επιληθούν στο εγγύς μέλλον. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας μαζί με το Κοινοβούλιο συνεργάζονται για να επιλύσουν το, τα θέματα, τα εκκρεμή ζητήματα στο εγγύς μέλλον. Υπάρχουν πολλοί τομείς ε, και πολλοί τρόποι επίλυσης και ελπίζω τα ζητήματα αυτά να επιληθούν στο εγγύς μέλλον έτσι ώστε να αρθούν όλα τα προσκόμματα για την Συμφωνία Σύνδεσης και την Συμφωνία Ελευθέρων Συναλλαγών. Τώρα, σε σχέση με θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας, εμείς θα προσχωρήσουμε στις συμβάσεις για την προστασία των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας. Δίνουμε τελική μορφή στη νομοθεσία μας για την προσέγγιση των νομοθεσιών και ότι συνδέεται ότι άπτεται θεμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας θα προσαρτηθεί στη Συμφωνία Ελευθέρων Συναλλαγών. Γι' αυτό θα Ήθελα να πω ότι πιστεύω ότι αυτό, ότι αυτό που σας ενδιαφέρει είναι οι, γεωγραφικές, οι γεωγραφικοί προσδιορισμοί, οι, οι γεωγραφικοί ορισμοί. Υπάρχει μια μεταβατική περίοδος, η κατονομασία των προϊόντων και ούτω καθεξής για να εξομαλυνθεί η κατάσταση. Σας ευχαριστώ πολύ. Λίγη το πρώτο τμήμα του workshop μας θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Κλούγεφ για τη συνεισφορά του, για την επιτυχία αυτής της συζήτησης. Σας ευχαριστώ και σας αποχαιρετώ. Now, let's move on. Ας προχωρήσουμε στο δεύτερο τμήμα της ε, συνεδρίασης. Ακούσαμε τους πολιτικούς. Ας ακούσουμε τώρα και τους εμπειρογνώμονες. Έχουμε επιφανείς εμπειρογνώμονες από την Πολωνία. Αναφέρομαι στον καθηγητή Μάρεκ Νταμπρόφσκι. Εκπροσωπεί το ΚΕΙΣ που είναι το Κέντρο για την ε, Κοινωνική και Οικονομική Ερεύνα στη Βαρσοβία. Κύριε Νταμπρόφσκι, έχετε διατελέσει υπουργό και βουλευτή ε, στην ε, Πολωνία. Είστε εμπειρογνώμονα για τα οικονομικά θέματα στην Ανατολική Ευρώπη. Ζήσατε χρόνια στην Ουκρανία και ήσασταν ε, Σύμβουλο για τα θέματα της ανατολική Εταιρικής Σχέσης επί σειρά ετών. Με αυτό το υπόβαθρο θα θέλαμε να ακούσουμε την ανάλυση σας σχετικά με τα διακυβεύματα της συμφωνίας αυτή. Έχετε το λόγο και σας ευχαριστούμε που ήρθατε. Καλώ ορίσατε. Thank you very much. Good morning. Ευχαριστώ και καλημέρα σε όλους. Θα ήθελα να ευχαριστήσω ε, την Επιτροπή Ίντεβ για τη σημερινή πρόσκληση. Είναι πάρα πολύ σημαντική και σχετικά ενδιαφέρουσα η σημερινή συνεδρίαση. Θα σας κάνω την παρουσίαση και υπάρχει ένα έγγραφο υποστηρικτικό ε, που συνέταξα ε, από κοινού με ένα συνεργάτη μου Θα ήθελα εξ αρχής ε, να σας πω ότι δεν πρόκειται για μία πρωτότυπη προσωμείωση για τους σκοπούς και τις ανάγκες της ε, συνεδρίασης. Δεν είχαμε αρκετό χρόνο στη διάθεσή μας ε, για να το κάνουμε αυτό. Έχουμε όμως εμπειρικά δεδομένα και άλλα στατιστικά δεδομένα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Ας αρχίσω με κάποια γεγονότα, δεδομένα σχετικά με τις εμπορικές σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ουκρανίας ε, και θα ήθελα να σας μιλήσω για την γενικότερη δομή ε, του εμπορίου στην Ουκρανία. Από πλευράς ε, εξαγωγών, ο Εθνικός Στατιστικός Οργανισμός της Ουκρανίας μας έχει δώσει συγκεκριμένα δεδομένα και βάσει αυτών είναι ο δεύτερος ε, εταίρος μετά την κοινοπολιτεία των εξαρτήτων κρατών από περιφερειακής ε, άποψης ε, και στο γράφημα βλέπετε ότι έχουν μειωθεί οι εισαγωγέ σε σχέση με την κοινοπολιτεία ανεξαρτήτων κρατών, αλλά προσοχή στην ερμηνεία, διότι αλλάζουν τα δεδομένα σε σχέση με τις διακυμάνσεις των ενεργειακών τιμών. Ε, και κατά τη διαστολή με τους πρώην ή τωρινούς υποψηφίους ή άλλους εμπορικούς εταίρους όπως ε, χώρες της ε, Βορείου Αφρικής θα διαπιστώσετε ότι είναι ο βασικός εταίρος της Ουκρανίας η Ευρωπαϊκή Ένωση από οικονομικής πλευράς ως εκ τούτου νομιμοποιούνται τα συμφέροντα της χώρας ε, και μπορούμε να ακολουθήσουμε και, ε, φυσικά και άλλες εμπορικές κατευθύνσεις από πλευράς Ουκρανίας σε σχέση με τη Ρωσία ή άλλες, ε, άλλα μέλη της κοινοπολιτείας ανεξαρτήτων κρατών. Επίσης με την Κίνα ε, από, οι εισαγωγές από την Κίνα αυξάνονται σταθερά. Θα, σχετικά τώρα με το δυναμικό της ε, Ουκρανίας ως προς εμπορικές σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση βλέπουμε ότι ε, ε, παρότι έχουμε επέλθει σε τέλμα σε σχέση με την αύξηση των εξαγωγών από τις αρχές του 2000 μέχρι το 2008, δηλαδή το τελευταίο έτος προκρίσης, οι εμπορικές ροές αυξήθηκαν ραγδαία περισσότερες ε, ε, εισαγωγές ε, προς την Ουκρανία και αντίστροφα. Ε, σημειώθηκε ραγδαία αύξηση λοιπόν. Το 2008 συρρυκνώθηκαν οι σχέσεις, ε, πλην όμως αυτό δεν είναι και κάτι που θα πρέπει να μας εκπλήσει, διότι ε, πρώτη φορά μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο συρρυκνώθηκε γενικότερα το διεθνές εμπόριο και μετά το 2009 παρατηρείται η ανάκαμψη. Όταν Εξετάζουμε την κατανομή ένα βασικό αγαθό ουσιαστικά για τις εξαγωγές. Ε, οι εξαγωγές ε, μεταλλευμάτων που περιέχουν σίδηρο ή όχι ε, υπερισχύουν στις εξαγωγές κατόπιν έχουμε πρώτες ύλες ή ημικατεργασμένα προϊόντα με μια κατηγορία πιο τελειοποιημένων αγαθών, συγκεκριμένα ηλεκτρονικά μηχανήματα που έχουν ε, από τις πιο σημαντικές θέσεις ε, στις εξαγωγές Επίσης, οι γεωργικές εξαγωγές έχουν κάποια σημασία, αλλά εδώ και είναι και η βασική διαφορά ανάμεσα στις εξαγωγές της Ουκρανίας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις εξαγωγές της Ουκρανίας ε, σε σχέση με άλλες γεωγραφικές κατευθύνσεις, ε, δηλαδή προς την κοινοπολιτεία ανεξαρτήτων κρατών και άλλες χώρες. Μέχρι στιγμής είναι σαφέστατο ότι οι γεωργικές εξαγωγές της Ουκρανίας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι κατώτερες, δεν έχουν ε, αξιοποιήσει το πλήρες δυναμικό. Αυτό σημαίνει ότι υπήρξαν σοβαροί εμπορικοί φραγμοί στο συγκεκριμένο τομέα. Σε σχέση με τις εισαγωγές από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ε, είναι πιο διαφοροποιημένα τα δεδομένα υπάρχουν υψηλότερε επενδύσει. Έχουμε δεδομένα από το 2010 και αν κάνουμε μία σύγκριση με το 2007 θα διαπιστώσουμε ότι τα μηχανήματα, ηλεκτρονικά μηχανήματα, ηλεκτρικά μηχανήματα κατέχουν την υψηλότερη θέση. Προφανέστατα με την κρίση συρρυκνώθηκαν οι επενδύσεις ε, και μειώθηκε η ζήτηση σχετικά με την, ε, τις αλλοδαπές επενδύσεις και σιγά σιγά αποκαθίσταται η τάση για αυτά τα ε, προϊόντα. Κατόπιν με τη συμφωνία αυτή την εις και σφαιρική συμφωνία ελευθέρων εμπορικών συναλλαγών DCFTA θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι στον οικονομικό στην οικονομία έχουμε διάφορους ορισμούς για αυτές τις συμφωνίες. Κάποιος ερευνητής ε, αναφέρθηκε ε, σε DCFTA και χρησιμοποίησε όρους όπως extensive DCFTA, δηλαδή εκτεταμένη και εις βάθος και σφαιρική συμφωνία. Τέλος πάντων δημιουργείται μια σύγχυση λόγω της ορολογίας. Ε, το θέμα, το ουσιαστικό θέμα είναι πως ε, υπάρχουν διαβαθμίσεις. Έχουμε συνολική ε, FTA, δηλαδή εμπορική συμφωνία, ε, συνολική κτλ. Αλλά αυτή η DCFTA, η σφαιρική συμφωνία, συνεπάγεται ότι πέρα από την κατάργηση των δασμών, Ε, υπάρχει και ένα ολοκληρωμένο θεματολόγιο για την μη δασμολογικών φραγμών, για την υιοθέτηση φυτοϊγειονομικών πρότυπων, κατάργηση τεχνικών φραγμών ε, στις εμπορικές συναλλαγές, που είναι και πολύ σημαντικές συνιστώσεις ε, τέτοιου είδους ε, συμφωνίας ε, για επίσης απελευθέρωση του εμπορίου για τις υπηρεσίες και κάτι άλλο που συνδέεται άρρηκτα με αυτό απελευθέρωση των επενδυτικών των διατάξεων περί επενδύσεων στην Ουκρανία και για να ολοκληρωθούν αυτοί οι στόχοι και να υλοποιηθούν αυτές οι συμφωνίες, οι υποφυσιολογικές συνθήκες ε, θα πρέπει να έχει προηγηθεί με ευρύτατη ρυθμιστική προσαρμογή μέσα από την ολοκλήρωση της ατζέντα σχετικά με την αμοιβή αναγνώριση. Η DCFTA, αυτή η εις συμφωνία υιοθετείται στα πλαίσια της ανατολικής εταιρικής σχέσης ε, και απορρέει, πηγάζει αν θέλετε από την Συμφωνία Εμπορίας ε, και Σύνδεσης ε, που υπέγραψε η Ευρωπαϊκή Ένωση τη δεκαετία του 90 με 10 νέα κράτη-μέλη που αναμένονται το 2004 και 7 να προσχωρήσουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κατόπιν ε, υπάρχουν αντίστοιχε συμφωνίες με υποψηφίου σε από τη Βαλκανική Χερσόνησο. Ε, ενιολογικά αποκομίσαμε ε, πλούσια εμπειρία από προηγούμενες ε, συμφωνίες. Ε, θα ήθελα τώρα να σας μιλήσω για τα αναμενόμενα ωφέλη και θα ήθελα να διηγηθώ, να ανατρέξω λίγο στο παρελθόν και στη συνέχεια να κάνω κάποιες εκτιμήσεις για το μέλλον. Θα ήθελα να αρχίσω από ε, διαπιστώσει κάποιων οικονομικών ε, μεγεθών. Ε, τα κέρδη και το κόστος της όδησης προς την υλοποίηση της συμφωνίας είναι υψηλότερο για την Ουκρανία σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί, διότι ε, μάλλον υπάρχει σειρά ε, λόγων, είναι ασύμε, υπάρχει ασυμμετρία ανάμεσα στους εμπορικούς εταίρους από πλευράς ε, οικονομικού δυναμικού και από πλευράς εμπορίου. στο πρώτο γράφημα που σας έδειξα νομίζω φαινόταν με σαφήνεια ότι το κομμάτι του του εξωτερικού εμπορίου της Ουκρανίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι κάτω από το 1 τρίτο τη Ευρωπαϊκή Ένωση προ την Ουκρανία και το αντίστοιχο τη Ουκρανία προ την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι στο 1%. Άρα υπάρχει ασυμμετρία ω προ το κόστο και ε, ω προ τα ωφέλη. Α ας με την Ουκρανία. Ε, καλύτερη πρόσβαση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πρώτα απ' όλα στην αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, σημαντικότατο ε, όφελος θα σας δείξω ε, στη συνέχεια. Επίσης μπορεί να εξυγχρονίσει την οικονομική της υποδομή η Ουκρανία και και από τις σημαντικότερες προκλήσεις. Απελευθέρωση των επενδυτικών καθεστώτων, σταθεροποίηση του επενδυτικού κλίματος. Αυτό σημαίνει μεγαλύτερη εισρωή αλλοδαπών επενδύσεων και Επίσης, ε, μεγαλύτερες ευκαιρίες να συμμετάσχει ε, στην παγκόσμια ε, αλυσίδα παραγωγής για τις βιομηχανικές εμπορικές συναλλαγές. Φυσικά, όπως προείπα, αναβαθμίζεται το επιχειρηματικό κλίμα, όπερ και έχει ιδιαίτερη σημασία για την Ουκρανία, γιατί στην αξιολόγηση της ε, ικανότητας ε, της Ουκρανίας ε, για συμμετοχή σε προγράμματα όπως το του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ της Παγκόσμιας Τράπεζας. Υπάρχουν διάφοροι διεθνείς δείκτες και ξέρετε ότι προς το παρόν η Ουκρανία δεν έχει καλή βαθμολογία. Ε, και η κατάσταση αυτή ε, δεν έχει βελτιωθεί τα τελευταία 50 χρόνια, οπότε ε, διακυβεύονται πολλά για την Ουκρανία. Η συμφωνία της EFTA ενδέχεται να βοηθήσει να βελτιωθεί η κατάσταση, αλλά είμαστε και ρεαλιστές. Ούτε η DCFTA, ούτε και η συμφωνία σύνδεσης δεν... Δεν είναι πανάκιες, και ε, υπάρχει και το οικονομικό σύστημα της Ουκρανίας όπου πρέπει να καταβληθούν εσωτερικές προσπάθειες για την εφαρμογή αυτής της συμφωνίας και για την πρόθεση αυτής της συμφωνίας. Τώρα όσον αφορά την Ευρωπαϊκή ε, Ένωση Ε, θα είναι πιο σταθερό το καθεστώς του εμπορίου και των επενδύσεων στην Ουκρανία για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης θα μπορέσει κανείς να επενδύσει στην οικονομική και πολιτική σταθερότητα της Ουκρανίας και να έχει πιο στενές σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και εδώ τώρα σας παρουσιάζω τα δυνητικά κέρδη από μια ευρεία FTA που διάφορες Προποθέσει προϋποθέσεις η οποία βασίζεται σε διάφορα ιστορικά στοιχεία δηλαδή καταρχήν μία πρώτη μελέτη της Γενικής Διευθύνσεως Εμπορίου του 2006 ε, η οποία βασιζόταν σε παλιά στοιχεία του 2001 ε, και βλέπουμε ε, τα ωφέλη για την Ευρώπη των 15 και λιγότερο για τα 10 κράτη που νέα κράτη-μέλη. Επίσης βλέπουμε μία αξιολόγηση για την ε, ε, Ουκρανία ε, η οποία είναι η πλέον εκτενής η οποία έχει γίνει στο θέμα αυτό βλέπουμε δε ότι από αυτές τις υπό αυτές τις προϋποθέσεις υπήρχαν αρνητικές βραχυπρόθεσμες ε, ε, αρνητικά βραχυπρόθεσμα κέρδη για την ευημερία της Ουκρανίας ε, της τάξης του μείων 5,29% και ουσιαστικά ε, βασιζόμαστε για τις προβολές αυτές σε παλιά στοιχεία της 2001, του 2004, του 2006, του 2007 ε, πριν από την κρίση στην, ε, στην παγκόσμια οικονομία και αυτό είναι επίσης ένας βασικός παράγοντας. Βλέπουμε λοιπόν ότι για την Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχουν πιο περιορισμένα αλλά σαφώς θετικά ωφέλη και πρέπει να προσπαθήσουμε να ε, βρούμε τα αποτελέσματα για τα μεμονωμένα κράτη-μέλη και να δούμε ποια από τα κράτη είναι αυτά τα οποία έχουν περισσότερες συναλλαγές αλλά και περισσότερα ωφέλη αλλά προς το παρόν όλα αυτά είναι υποθέσεις. Τώρα, οι, οι επιπτώσεις ανατομέα που βασίζονται σε, ε, στις στατιστικές. Βλέπουμε ότι υπάρχει μία πιο ο, νέα κατάσταση και βλέπουμε ότι ε, σε ορισμένους τομείς στην Ουκρανία όπως είναι η μεταλλουργία, ε, η μεταποίηση, τα, ε, η κλωστοεφαντουργία υπάρχουν γενικώ ωφέλη που διαπιστώνονται και εδώ πρόκειται για μια μελέτη του 2007 όπου λέγεται ότι θα υπάρχουν ωφέλη για την Ουκρανία στην ορυκτή παραγωγή, στα κρέατα ή στη ζάχαρη, στον μεταφορικό εξοπλισμό και στις ε, ε, οικονομικές υπηρεσίες. Δεν είναι τόσο σαφής η κατάσταση ενώ για την Ευρωπαϊκή Ένωση ουσιαστικά θα ωφεληθεί η βιομηχανία Τώρα μιλούμε ε, για διάφορες διαπραγματεύσεις. Πρέπει ε, να πούμε ότι δεν υπάρχει πληροφόρηση του κοινού σχετικά με το DCFTA ε, το περιεχόμενο και τις λεπτομέρειες των διαπραγματεύσεων ε, σχετικά με τα πιο σημαντικά θέματα από ό,τι γνωρίζουμε το προ σημαντικό θα είναι το μέγεθος των δασμολογικών ποσοστώσεων για τις ε, γεωργικές εισαγωγές από την Ουκρανία επίσης η προστασία εισαγωγών για την ε, αυτοκινητοβιομηχανία στην Ουκρανία, η κατάργηση των εξαγωγικών ε, ε, δασμών στην Ουκρανία που αναφέρθηκε και σήμερα, η προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων στην Ουκρατία, το εμπόριο και η συνεργασία στον ενεργειακό τομέα και η ελεύθερη πρόσβαση στην ευρωπαϊκή αγορά για τις υπηρεσίες μεταφορών δεν έχω χρόνο για να σχολιάσω αυτά τα θέματα αλλά πιστεύω ότι δεν υπάρχουν ε, τόσα πολλά αμφιλεγόμενα θέματα και ότι θα μπορέσουμε ε, να ε, καλύψουμε τις βασικές προϋποθέσεις και πέραν αυτού ότι θα ε, μπορέσουμε να ε, αντεπεξέλθουμε αυτών των διαπραγματεύσεων. Αυτό όμως που είναι κρίσιμο ε, για να μπορέσει να ολοκληρωθεί η συμφωνία αυτή είναι η ανησυχία της Ευρωπαϊκής Ενώσεως σχετικά με τις πολιτικές ελευθερίες, τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου στην Ουκρανία. Δεν υπάρχει κίνδυνος κυρώσεως από την πλευρά της Ουκρανίας, αλλά υπάρχουν σοβαροί κίνδυνοι που αναφέρονται στην ανεπαρκή εφαρμογή εφαρμογή του DCFTA ε, από ουκρανικής πλευράς και πολιτικής και Κοιτικής. Ε, ξέρουμε ότι το κυβερνών κόμμα είναι υπέρ αυτής της συμφωνίας, παραμένουν όμως ε, οι κίνδυνοι για την εφαρμογή αυτής της συμφωνίας στην Ουκρανία και τα προβλήματα τα οποία έχουν προκύψει επανειλημμένως στο παρελθόν μπορεί να ξαναπροκύψουν και τώρα δηλαδή η ε, πρόσβαση και η εφαρμογή των υποχρεώσεων του ΠΟΕ ε, τα θέματα που έχουν σχέση με την ε, ικανότητα εφαρμογής ε, διότι ε, βλέπουμε ότι υπάρχει ενδιαφέρον και υπάρχει και η κριτική και η κρίσιμη νομοθεσία η οποία όχι μόνο θα πρέπει να ψηφιστεί αλλά και να εφαρμοστεί. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ για αυτήν την, την παρουσίαση. Ε, τα δεδομένα αυτά θα είναι διαθέσιμα προς το κοινό όταν θα είναι έτοιμα τα πρακτικά της συνεδρίασης. Very... Αυτό που έχει σημασία είναι να λάβουμε υπόψη τους έγκριτους ε, προσκεκλημένους μας, διότι συμμετείχα στις διαπραγματεύσεις. Μιλώ για τον κύριο Πίτερ Μπάλας, που είναι Γενικός Διευθυντής στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Γενική Διεύθυνση Trade, και τον κύριο Πιανίτσκι, ο οποίος είναι Υπουργός Οικονομίας. Από όσο κατανοώ υπάρχουν ε, ορισμένοι περιορισμοί. Δεν μπορούν δηλαδή να μας μιλήσουν για το περιεχόμενο, το πλήρες περιεχόμενο της συμφωνίας, διότι πρώτα θα πρέπει να δοθούν αυτά τα στοιχεία στα δύο κράτη και στα μέλη του Κοινοβουλίου. Μπορείτε ίσως να μας πείτε για τα βασικά ζητήματα στα οποία αναφέρθηκε ο κύριος Τραμπόφσκι. Ο Πίτερ Πάλας έχει το λόγο, που είναι και πάλι μαζί μας. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Θα ήθελα και εγώ να εκφράσω τις ευχαριστίες μας προς τον καθηγητή Νταμπρόφσκι, διότι πραγματικά μας έδωσε πολύτιμα στοιχεία για να αναλύσουμε την κατάσταση. Θα ήθελα όμως να κάνω δύο σχόλια. Σε σχέση με αυτά που είπε ο Πρόεδρος, όπως ακούσατε, βασικά ζητήματα των διαπραγματεύσεων ολοκληρώθηκαν χτες το βράδυ και υπάρχουν εκρεμή νομοθετικά ζητήματα, τα οποία επιλύονται τώρα. Γιατί αυτό που έχει σημασία είναι να ειδωθεί το κείμενο από τα δύο από, την Ουκρανία και από τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ο καθηγητής Νταμπρόφσκι μας είπε ότι δεν έχουμε λεπτομέρειες διαθέσιμες, δηλαδή συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις, τίποτα δεν έχει συμφωνηθεί, δεν μπορούμε να πούμε ότι έχει συμφωνηθεί παρά όταν έχουμε ολοκληρωμένη συμφωνία. Δεν θέλουμε λοιπόν να συμμεριστούμε αυτές τις λεπτομέρειες, διότι δεν ξέρουμε ποια θα είναι η έκβαση των συζητήσεων. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί λοιπόν και να δούμε τις πληροφορίες που έχουμε στη διάθεσή μας μαζί με το Κοινοβούλιο και να μπορέσουμε να δούμε ποιες είναι και οι λεπτομέρειες. Ένα άλλο στοιχείο είναι ότι εξ αρχής, από την αρχή των διαπραγματεύσεων, ε, παρευρέθηκα στις συναντήσεις και θα πρέπει να αναφερθώ στον Ρούπερτ Σλέγκερ, ο οποίος συμμετείχε στο τελικό στάδιο των διαπραγματεύσεων. Ε, είναι μαζί μας από την Γενική Διεύθυνση Τρέν, λοιπόν. Θα ήθελα να κάνω ορισμένα σχόλια και εγώ θα ήθελα να πω ότι αυτή η DCFTA είναι ένα, είδο, ένα ε, νέο είδος συμφωνίας που μέχρι τώρα δεν είχε υπογραφεί με καμία άλλη χώρα. Η Ουκρανία θα είναι η πρώτη. Ελπίζουμε οι συμφωνίες να φτάσουν σε αίσιο πέρας και υπάρχουν ορισμένες ομοιότητες με τις προγενέστερες συμφωνίες σύνδεσης, αλλά υπάρχουν και ορισμένες διαφοροποιήσεις που σχετίζονται με την ίδια τη φύση της συμφωνίας ε, σύνδεσης, ιδιαίτερα ως προς την πλαισίωσή της. Όταν όμως δούμε την DCFTA, αυτή τη σφαιρική και σε βάθος συμφωνία ελευθέρων συναλλαγών, μιλάμε για υψηλή ολοκλήρωση και βλέπουμε ότι η Ουκρανία προσχωρά εμπολής στην εσωτερική αγορά. Δεν πρόκειται βεβαίως για συμφωνία σύνδεσης καθεύτη. Γι' αυτό υπάρχουν ορισμένα στοιχεία όπως η ελεύθερη κυκλοφορία γεωργικών αγαθών που δεν προβλέπεται από αυτή τη συμφωνία και η ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων. Άρα αυτό έχει σημασία με τις τέσσερις βασικές ελευθερίες, αλλά σε αυτά τα ε, πλαίσια και αυτό που έχει σημασία είναι η ολοκλήρωση όπως προβλέπετε, έτσι ώστε βαθμιδών να ισχύσει. Είναι πολύ ε, ενδιαφέροντα αυτά τα επιμέρους ζητήματα, διότι ακόμα και αν δεν ισχύουν αυτά τα στοιχεία που είπε ο συνάδελφος, Μιλάμε τουλάχιστον ε, για ε, δέκα νέα δεδομένα μεταξύ Ουκρανίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης και αν θέλουμε να είμαστε ακριβείς υπάρχουν ε, περιορισμοί στην πρόσβαση στις αγορές. Εσείς αναφερθήκατε στη γεωργία ως προς τα ευαίσθητα αγωθά θα υπάρξουν δασμολογικές απελευθερώσεις αλλά και περιορισμοί, αλλά νέες δυνατότητες εξαγωγών. Είδαμε για, μιλήσαμε για μια τάξη του 4 έως 7% δασμολογικές ελαφρύνσεις Η Πολωνία έχει πολλά να κερδίσει από αυτή τη συμφωνία, δηλαδή γενικά οι γείτονες χώρες. Και θα είναι μεγάλη όθηση και για την ανάπτυξη των δύο πλευρών. Ευχαριστώ. Ας ακούσουμε την άποψη της ουκρανικής πλευράς, ο κύριος Πιατνίτσκι, ο οποίος είναι αναπληρωτής υπουργός οικονομικών της χώρας. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Αγαπητοί, αγαπητά μέλη, είχαμε πολύ ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Ντομπρόσκι για αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίαση. Ακούσαμε για πολλά στοιχεία, αριθμητικά στοιχεία ως προς το εμπόριό μας με την Ευρωπαϊκή Ένωση και από όσο, από μιλάμε για έρευνες οι οποίες περιλαμβάνουν πολλά επιμέρους στοιχεία. Αυτό που έχει σημασία είναι να δούμε πώς αναπτύχθηκε, πώς αναπτύχθηκε αυτό το εμπόριο. Ποιο είναι το ιστορικό. Αλλά δεν μπορούμε να μιλήσουμε μόνο για το ιστορικό σκέλος, δηλαδή αυτό που οδήγησε στην ανάπτυξη των σχέσεων μπορώ να σας αναφερθώ σε ορισμένους παράγοντες που υπησύλθαν και προώθησαν τις εμπορικές μας σχέσεις. Ελπίζω αυτοί οι παράγοντες να ειδωθούν και να αντιμετωπιστούν σωστά. Βεβαίως η Ουκρανία μετά την ε, ανεξαρτησία της και αφού αποχώρησε από την πρώην Σοβιετική Ένωση ε, έζησε μία περίοδο οικονομικών και πολιτικών κλειδονισμών. Άρα στην αρχή της ανεξαρτησίας μας είχαμε πολλές προκλήσεις να αντιμετωπίσουμε, μέτρα dumping και άλλα μέτρα προστατευτισμού. Και βεβαίως τα αγαθά μας δεν υπησέρχονταν και δεν λαμβάνονταν υπόψη στην ευρωπαϊκή αγορά. Τώρα μας φαίνεται περίεργο όταν κοιτάμε προς τα πίσω και βλέπουμε τα μέτρα που ακόμα ισχύουν και που εισήχθησαν το 98-99 προϊόντα μεταλλουργίας, χημικά και όπως είπα ήδη μεταλλουργίας για σωληνώσεις μιλάμε για δεκάδες εκατοντάδες δολάρια, προϊόντα που ακόμα δεν, είχαν, δεν έχουν πρόσβαση, δεν μπορούν να μπουν στις ευρωπαϊκές αγορές και θα πρέπει να πούμε ότι από ευρωπαϊκής πλευράς θα φτάσουμε στην πλήρη απελευθέρωση. Αλλά το 52% ε- των δασμών που αφορούν τα προϊόντα μεταλλουργίας υπησέρχονται στα μέτρα αντι-dumping. Άρα κατανοούμε ότι αυτά τα αγαθά δεν θα φτάσουν στις ευρωπαϊκές αγορές και οι δασμοί που ανέρχονται σε ένα 52%. Αυτός ο δασμός του 52% ίσχυε το 98%. Γιατί μιλάμε λοιπόν. Μπορούμε να μιλήσουμε περισσότερο και για την διαδικασία διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2004, όπου αλλάξαν τα δεδομένα με αυτή τη διεύρυνση. Δέκα νέε χώρες προσχώρησαν στις δομές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και φτάσαμε σε μία συμφωνία όπου λάβαμε κάτι κάτω από το ίμιση των προμηθειών μας από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα Εμείς προμηθεύσαμε την Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή προωθήσαμε τα προϊόντα μας, αλλά οι προμήθειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έπεσαν κατά το ίμιση μετά από αυτή τη νέα προσχώρηση του 2004. Ίσως το πεδίο εφαρμογής των εμπορικών συναλλαγών δεν είναι τόσο ευρύ όσο θα επιθυμούσαμε. Αλλά αυτό που έχει σημασία είναι ότι υπάρχει μία διεύρυνση ως προς την εξαγωγή ορισμένων αγαθών. Θα θέλαμε όμως στο μέλλον να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα και όταν αναλύσουμε τα ευεργετήματα κατανοούμε ότι αυτή η συμφωνία είναι ύψης της σημασίας. Μιλήσατε για την βιομηχανία ζάχαρης, για τη μεταποιητική βιομηχανία. Αυτό που μας ενδιαφέρουν είναι τα ευεργετήματα. Εσείς μιλήσατε για ποσοστώσεις, αλλά είναι δύο φορές μικρότερη αυτή η ποσόστοση από την αρχικά προβλεπόμενη. Αυτό που έχει σημασία λοιπόν είναι να δούμε τα μεγέθη. Μιλάμε για πολύ διαφορετικά μεγέθη ως προς την κατεργασία ζάχαρης. Γι' αυτό εμείς ε, ανοίγουμε τις αγορές μας για να φτάσουμε σε μηδενικούς δασμούς, τουλάχιστον ως προς τη ζάχαρη. Ελπίζουμε να απελευθερωθεί η κατάσταση και σε άλλους τομείς, αλλά πολλές φορές οι εταίροι μας δεν είναι έτοιμοι. Θα πρέπει να δούμε ποια συνέχεια θα δοθεί ποιες είναι οι μελλοντικές προοπτικές ως προς τη γεωργία σήμερα, διότι σήμερα δεν ξέρουμε τι θα γίνει με τους δασμούς σε 5, 10, 15 χρόνια. Υπάρχουν ακόμα δασμοί. Τι θα γίνει όμως βαθμιδών. από πλευράς Ουκρανίας η διαδικασία απελευθέρωσης βρίσκεται εντογίγνεσθε, πρόκειται για μια διαφανή διαδικασία και αυτό το κατανοούν οι επιχειρήσεις. Στην Ευρώπη όμως τι θα γίνει. Θα υπάρχει ανταπόκριση. Άρα βλέπουμε ότι δεν υπάρχουν μόνο αρνητικά στοιχεία. Όταν αναλύσουμε όμως τις διαδικασίες, τις εξελικτικές αυτές διαδικασίες μας ενδιαφέρει να δούμε κατά πόσο υπάρχει σαφήνεια και ευκρίνεια. Όταν μιλάμε για προϊόντα κρέατος, για το κρέας θα πρέπει να ακολουθήσουμε τις προπετήσεις που υπάρχουν ως προς τον ε, τις υγειονομικές προδιαγραφές. Αν όμως ε, γίνουν έρευνες θα πρέπει να δούμε κατά πόσο υπάρχει προσέγγιση νομοθεσιών και κατά πόσο οι δικοί μας εταίροι θα μπορούσαν να έχουν πρόσβαση στην αγορά. Γιατί δεν μπορούμε να έχουμε μια διαφορετική προσέγγιση σε σχέση με τη Ρωσία ή την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμείς θα προσεγγίσουμε πολύ περισσότερο την ευρωπαϊκή αγορά. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την προσοχή σας και αν υπάρχουν ερωτήσεις είμαι έτοιμος να απαντήσω. Πριν δώσω το λόγο στο... Ζητήσω από τον καθηγητή Νταμπρόσκι να πάρει το λόγο για αυτό το δεύτερο τμήμα της συνεδρίασης. Ε, θα ήθελα να δω αν υπάρχουν ερωτήσεις. Ε, από τα... Ας αρχίσουμε με τους βουλευτές της Επιτροπής ΙΝΤΕ. No questions. Δεν υπάρχει καμία ερώτηση. Ε, φαίνεται ότι είναι σαφέστατα όλα. Έχετε κύριε Νταμπρόφσκι κάποια καταληκτικά σχόλια. Έχετε κάτι να προσθέσετε στις, ε, ε, στην πρώτη σας παρουσίαση. Ευχαριστώ. Καταλαβαίνω για ποιο λόγο το περιεχόμενο της συμφωνίας και οι λεπτομέρειες ε, των διαπραγματεύσεων ε, ε, μπορούν να οδηγήσουν μόνο σε διαπιστώσεις δεν μπορούμε λοιπόν πλήρως να βασιστούμε σε αυτά. Θα ήθελα να ε, συμφωνίζω με ε, τον προλαλήσαντα και να σχολιάσω και κάτι που ακούστηκε εδώ κατά τη διάρκεια της συζήτησης. Η κοινή γεωργική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν θα μεταρρυθμιστεί άρδιν ε, υποφυσιολογικές συνθήκες και αυτό θα θέσει σημαντικούς περιορισμούς στην συμφωνία Στι διαπραγματεύσει για σύναψη εμπορικών συμφωνιών με τους διάφορους εταίρους Ευρωπαϊκής Ένωση. Ε, Παραδείγματο χάρη ένα από του συντάκτε ε, τη έρευνας ε, που σας έλεγα προηγουμένως, δεν πρόλαβα, δεν πρόλαβα να το σχολιάσω την πρώτη μου παρέμβαση αυτό, τέλος πάντων, ένας από τους συντάκτε έκανε ένα παραλληλισμό με την επερχόμενη συμφωνία με τη Γεωργία ε, διακόπτει ο πρόεδρος, ο κύριος Μορέιρα. Μπορείτε θέλετε λίγα λεπτά για να προετοιμαστείτε και να μας το παρουσιάσετε αυτό το σημείο. Αν θέλετε λεπτομέρειες, ναι, δύο-τρία λεπτάκια. Δεν χρειάζεται, απαντάει ο κύριος ε, Νταμπρόφσκι. Η Γεωργία και η Μολδαβία έχουν θεσμικές και οικονομικές ε, συνάφειες, ε, μάλλον ε, ομοιότητες με την Ουκρανία, γιατί ήταν όλες πρώην Σοβιετικές δημοκρατίες. Ως προς το μέγεθος της οικονομίας όμως και ως προς τη δομή της οικονομίας υπάρχουν σημαντικές διαφορές. Υπάρχει, είναι πιο γεωργικές οικονομίες ή βασίζονται περισσότερο στις υπηρεσίες και όχι τόσο στα αγαθά. και θεωρώ ότι θα ανακύψουν λιγότερε δυσκολίε κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων σχετικά με την προστασία κάποιων βιομηχανικών ε, συμφερόντων. Αλλά το θέμα που έθιξε ο κ. Πιατνίτσκι σχετικά με την προοπτική των αγροτικών εξαγών προ την Ευρωπαϊκή Ένωση θα έχουν ακόμη μεγαλύτερη σημασία. Για την Μολδαβία που εξάγει λαχανικά και κρασιά και το ίδιο και για τη Γεωργία είναι θεμελιώδε το ζήτημα. Και το ίδιο για την εξαγωγή εργασίας ε, και υπηρεσιών, άρα και ελεύθερη κυκλοφορία των ε, προσώπων. Ε, ως προς το ΑΕΠ τα εμβάσματα στην ε, Μολδαβία δυστυχούσαν ε, σε πάνω από 7% του ΑΕΠ. Όχι ότι δεν είναι σημαντικό αυτό για την Ουκρανία, αλλά όχι τόσο σημαντικό όσο για τη Μολδαβία. Άρα υπάρχουν διαφορές ανάμεσα στις δύο οικονομίες. Σχετικά τώρα με το εμπόριο των γεωργικών προϊόντων, με την ιδιότητα του εμπειρογνώμων, αντιλαμβάνομαι γιατί υπάρχουν διάφοροι περιορισμοί σε αυτό το τομέα και σκεφτείτε και τη, ταυτόχρονα και τι διαπραγματεύσει ε, στα πλαίσια του ΠΟΕΣ τη αλλά για λιγότερο ανεπτυγμένε χώρες ε, ε, και ας μπούμε τώρα στο πλαίσιο της ανατολικής εταιρικής σχέσης υπάρχουν χώρες και υπάρχουν ανατολικοί γείτονες και νότιοι γείτονες για τους οποίους αυτά τα ζητήματα έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα. Αφενός Αντιλαμβάνομαι ότι θέλετε να κάνετε παραλληλισμό με άλλες εμπορικές ε, συμφωνίες, διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση τώρα έχει την πρόθεση να προχωρήσει περισσότερο σε σχέση με το παρελθόν. Π.χ. αν συγκρίνουμε με την εμπορική συμφωνία με ε, νότιες χώρες ε, της Μεσογείου τη δεκαετία του 90, τώρα λοιπόν προτίθεται να προχωρήσει την περαιτέρω η Ένωση και ο κ. Πιατνίτσκι νομίζω είχε τα σωστά ζητήματα, διότι το κόστος προσαρμογής για κάποιους συγκεκριμένους παραγωγούς στα, στις χώρες εταίρους της Ένωσης είναι σε ιδιαίτερα ψηλά επίπεδα, μιλώντας για υιοθέτηση φυτογειονομικών ε, προτύπων, ποιοτικών προτύπων κτλ. Οι πρόπτικες, ε, λοιπόν είναι συγκεκριμένες. Ε, πώς ακριβώς θα καταργηθούν οι ποσοστώσεις τα επόμενα 15 χρόνια. Είναι σοβαρότατο αυτό το πρόβλημα. Είναι λογικό ε, ε, να αναλάβουμε τέτοιο κόστος, τέτοιο υψηλό κόστος προσαρμογής, αναρωτιέται κανείς και δικαίως. Ε, και νομίζω ότι οι προσπάθειες θα πρέπει να γίνονται αμφωτέρων των πλευρών. Αυτό είναι το καταληκτικό μου σχόλιο. Πρόεδρος, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και φτάνουμε στο τέλος ε, των εργασιών μας, ε, αλλά ο κύριος Πάβελ Ζαλεύσκη, που είναι ο μόνιμος εισηγητής μας, θα πάρει το λόγο για να κάνει κάποιες καταληκτικές παρατηρήσεις και να αντλήσει τα συμπεράσματα της συζήτησης. Uh, Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και για την προσωπική σας συμμετοχή σε αυτή την εργασία, διότι πιστεύω ότι όλοι γνωρίζουν πόσο σημαντικό ήταν να παρουσιαστούν όλα αυτά τα θέματα και να αυξηθεί η συνειδητοποίηση στο Κοινοβούλιο ότι ε, πρέπει να γνωρίζουν όλοι πόσο σημαντική είναι αυτή η συμφωνία CDFTA. Δεν φτάνει να, είναι, να έχει κανείς δίκιο αλλά να έχει δίκιο την κατάλληλη στιγμή. Ε, νομίζω ότι αυτό έχει αποδεικτεί στην ιστορία αυτής της Επιτροπής και ε, συνήθως ε, η ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων ανακοινώνεται. Είναι δηλαδή ένα βασικό πολιτικό μήνυμα το οποίο πρέπει να περάσει. Όλοι τόνισαν πόσο σημαντικό είναι όχι μόνο από οικονομικής απόψεως πράγμα το οποίο είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικό να μπορέσει να ε, ενταχθεί η ε, ουκρανική οικονομία στην ε, ευρωπαϊκή και πρέπει όλοι να μπορούν να εφαρμόσουν αυτή τη συμφωνία. Η προοπτική ουσιαστικά είναι να δημιουργηθεί ε, μία σταθερή μεγάλη χώρα ε, και με τις νέες εξελίξεις θα μπορέσει να αποτελέσει μέρος της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και αυτή η χώρα. Ε, είχαμε λοιπόν ένα καλό πρότυπο με την ε, Πολωνία που είναι επίσης μια μεγάλη χώρα με την οποία έγινε μία συμφωνία ελευθέρω εμπορίου το 92 ε, και μετά προσχώρησε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τώρα το ΑΕΠ είναι πολλαπλάσιο της Ουκρανίας. Είναι λοιπόν μια απόδειξη για το πόσο σημαντικό είναι να εφαρμόσει κανείς σωστά αυτή τη συμφωνία και ε, νομίζω ότι συζητήσαμε για την πολιτική πτυχή αυτής της συμφωνίας αλλά είναι πολύ σημαντικό και συμφωνώ με αυτό το οποίο είπε ο, ο, Επίτροπος και ο εκπρόσωπος της Πολωνικής Προεδρίας. Εδώ όμως μιλούμε για το μέλλον περίπου 50 εκατομμυρίων ατόμων. Μιλάμε για αλλαγή πολιτισμική και για ε, την διαμόρφωση της, ε, του εσωτερικού ειδικού πολιτικού προγράμματος της ε, Ευρώπης, της ε, Ουκρανίας που θα πρέπει να προσαρμοστεί στην Ευρώπη μέσω της εφαρμογής αυτής της συμφωνίας συνδέσεως και του TFTA. Και τέλος θέλω να σας πω και αυτό είναι η παράκλησή μου προς την Επιτροπή ότι θα μπορέσουμε μετά να ε, την εφαρμόσουμε ε, σαν ε, προσωρινή συμφωνία δηλαδή να μην διστάσουμε, να μην χρονοτριβήσουμε και να την εφαρμόσουμε αμέσω. Ευχαριστώ. Φαντάζομαι ότι όλοι συμφωνείτε ότι αυτή η, η συζήτηση ήταν πάρα πολύ επικοδομητική και ιδίως σχετικά με την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων και για την εξαιρετική ποιότητα των ομιλητών οι οποίοι μπόρεσαν να μας ενημερώσουν σχετικά με ε, αυτήν την σημαντική συμφωνία διότι ξέρετε ότι το Κοινοβούλιο με βάση τις τη της Λισαβόνας έχει δικαίωμα όχι μόνο να ακυρώνει τις συμφωνίες αλλά να ενημερώνεται και να συμμετέχει στις διαπραγματεύσεις οπότε καλό είναι να γνωρίζουμε ε, τα διακυβδέματα αυτής της συνεργασίας και πρέπει να σας πω ότι κατά τη γνώμη μου αυτή ήταν ε, μια πολύ καλή στιγμή της ε, κοινοβουλευτικής ε, δημοκρατίας. Ευχαριστώ και την Γραμματεία και την Πολιτική Επιτροπή που ετοίμασαν αυτή την συνεδρίαση και τέλος όλους από εσά που ήρθαν και συμμετείχαν σε αυτήν την συνεδρίαση. Και τέλος, μία τελευταία παρατήρηση το πρωτόκολλο ασφαλείας απαιτεί να ακολουθήσουμε τους φιλοξενούς μας μέχρι την είσοδο του Κοινοβουλίου. Σας παρακαλώ λοιπόν να εντοπίσετε τους υπευθύνους έξω από την αίθουσα που θα σας οδηγήσουν προς την έξοδο. Σας ευχαριστώ.